πρακτικά. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων στην ε, συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου ενέκρινε τις ε, εντολές τριών συναδέλφων και ζητάει από την Ολομή να κάνει το ίδιο. Πρόκειται για τον κύριο Ινιάκη Μπαλμπέιτα Φερνάντες από 11 Ιουλίου, τον κύριο Εντουάρτ Ραούλ Χέλβιχ και τον κύριο Οβίδιου Ιωάνν Σιλάγη από 4 Σεπτεμβρίου και για την κυρία Μαρτίνα Μίχελς από 5 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει κάποια αντίρρηση? Οπότε εγκρίνονται οι εντολές των συναδελφών. Η κυρία Νέσα Τσάλτερς Τσίλτερς